για την κατάσταση βίας κατά των γυναικών στην Ινδία. Υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων και του κυρίου Πάσκα που μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ψήφισμα. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκέκρινται ομόφωνα το, κοινό ψήφισμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Έχουμε μετά άλλα έξι ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαχρέιν. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα των έξι κομμάτων και του κυρίου Πάσκα. Και έχουμε μια προφορική τροποποίηση για την παράγραφο 10 της κυρίας Ανδρίκηνα. Κύριε Πρόεδρε, Εξ ονόματος της του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω αυτή την προφορική τροποποίηση για την παράγραφο 10. Και είναι μονάχα μια λέξη. Η λέξη άμεσα. Επομένω η παράγραφο 10 θα λέει υπογραμμίζει την ισχυρή ε, έλλειψη υποστήριξη για την έλλειψη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση των Παχρέν ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να καταδικάσει τι συνεχιζόμενε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και να εφαρμόσει στοχευμένε κυρώσει απαγορεύσει βίζα και πάγωμα στοιχείων ενεργητικών εναντίον των ατόμων αυτών που είναι άμεσα, και εδώ είναι η τροποποίηση, άμεσα εμπλέκονται στι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Όπω αναφέρεται στην έκθεση του BICI, και να επανεξετάσει τι σχέσει σε ε, διπλωματικό και εμπορικό επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Μπαχρέιν. τέλο τη παράθεση. Ευχαριστώ κυρία Αντρίκενα. Υπάρχουν αντιρρήσεις κατά της προφορικής αυτής ε, τροποποίησης. Όχι. Ψηφίζουμε την παράγραφο 10 σε δύο τμήματα. Ένα πρώτο τμήμα με την λέξη directly, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, γίνεται δεκτή αυτή η τροποποίηση. Το υπόλοιπο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται το δεύτερο αυτό τμήμα. Ερχόμαστε στο ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί, ψήφι υπέρ, κατά αποχές και ομόφωνα εγκρίνεται και αυτό το ψήφισμα και ερχόμαστε στο, στα έξι ψηφίσματα για την κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία και εδώ έχουμε ένα κοινό ψήφισμα έξι κομμάτων και του κυρίου Πάσκα δεν υπάρχουν τροπολογίες ψηφίσουμε στο σύνολο το ψήφισμα αυτό με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Με 51 ψήφους υπέρ και μία αποχή εγκρίνεται η, το ψήφισμα αυτό το κοινό. Τα πρακτικά τη ε, συνεδρία αυτή θα δοθούν για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους αποδέκτες τους. Η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διακοπεί και σας εύχομαι σε όλους καλή και ασφαλή επιστροφή και ωραίο Σαββατοκύριακο.